Pa Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah, Mr. Borelli is not here, so we start with your... Ο κύριος Μπορέλη δεν είναι εδώ, ήρθε θα ξεκινήσουμε με τον Παύλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν γνώριζα ότι είναι το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την τελευταία μα συνεδρίαση σκέφτηκα περαιτέρω τη συμφωνία και θέματα που θέλω να συμπεριλάβω στην έκθεση μου. Έλαβα υπόψη κάποιες ιδέες ε, που εξέθεσε η Επιτροπή Ντεβ στην γνωμοδότησή της και επίσης ε, ζήτησα και με τους ε, σκιώδες ηγητές. Το πρώτο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι πιστεύω ότι το Trade Facilitation Agreement είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Θα βοηθήσει την εισαγωγή προϊόντων ε, με πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με την, καθυστέρηση, με την αποφυγή καθυστερήσεων στα σύνορα. Αυτό είναι πολύ καλό για τις υποανάπτυξη χώρες έτσι τους δοθεί τεχνολογική ε, βοήθεια για να εξχρονίσουν τι τελειωνικές διαδικασίε Επιπλέον αυτό αποτελεί καλή είδηση για την πολυμερή ατζέντα γιατί δείχνει ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μπορεί να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι σύμφωνα με τι συνθήκες του 21 ου αιώνα και γι' αυτό προτείνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη συνέντευξή του σε αυτή τη συμφωνία. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ε, σημεία στο σχέδιο έκθεσή θέλω να τονίσω κάποια από αυτά. Πρώτα απ' όλα, τα ωφέλη της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας ε, έχουν γίνει μελέτες από αυτού για να μετρήσουν ε, τις επιπτώσεις και να είναι σαφές ότι αυτή η πολύ σημαντική συμφωνία θα μπορέσει να μειώσει το κόστος ε, του εμπορίου κατά 10%, περισσότερο από 10%, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για την πρόσβαση σε νέες αγορές. Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι ε, το εξής. Θα ήθελα να είναι σημαντικό προς την ανάπτυξη αυτή η συμφωνία. Θα διδοθούν πολλά κονδύλια για, την, για να βοηθούν η παράπτυξη και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Θα υπάρξουν και μεταβατικές περίοδοι και, ε, και οικοδόμηση ικανότητων φυσικά. Θα ήθελα επίσης να τονίσω κατά τρίτον το συντονισμό. Υπάρχουν ε, πολλοί εμπλεκόμενοι, ο ΠΟΕ, ο ΣΑ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων. Ο συντονισμός και η συνεργασία αποτελεί κλειδί ώστε η χρηματοδότηση και η πυρογνωσύνη να ε, πάει εκεί που ακριβώ χρειάζεται, ώστε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Τέλος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Θα ήθελα να υπάρξει επικύρωση στην πλευρά του ΠΟΕ ώστε να υπάρξει να είναι ήδη σε εφαρμογή ε, πριν από την σύνοδο που θα γίνει στο Ευρώπη το Δεκέμβριο. Και χρειάζεται μια συγκεκριμένη πλειοψηφία στην ψηφοφορία. Θα πρέπει εδώ στο Κοινοβούλιο να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή ένιση αντιστοιχεί σε 20 ψήφους στον ΠΟΕ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου και προσβλέπω στην υποστήριξη των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πάμπλο. Τώρα η σειρά στους σκιώδεις εισηγητές κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή για το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο γνωμοδότησης που είναι λεπτομερές και που τονίζει τη σημασία αυτή τη συμφωνία, γιατί είναι μια πολυμερή ε, συμφωνία. Κατά δεύτερον, επειδή είναι μια συμφωνία που, όπω ε, είπε ο εισηγητή, μειώνει τα έξοδα της δαπάνης του παγκόσμιου εμπορίου. Και θα δώσει παράλληλα μεγάλες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί το διοικητικό κόστος θα μειωθεί. και θα υπάρξουν πολλές διευκολύνσεις. Είναι καινοτόμο συμφωνία η οποία θα είναι ε, στα μέτρα των συγκεκριμένων χωρών και που θα επιτρέψει ακόμα και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να λάβουν τεχνική υποστήριξη. Ε, βοήθεια από τις χώρες δωρητές και να έχουν τους πόρους για την εφαρμογή της συμφωνίας ακόμα και στις λιγότερο πραγμανές χώρες όπου ο τεχνικός μηχανισμός δεν είναι τόσο παρκής να τονίσει κάποια άλλα σημεία χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία έχουμε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων στον ΠΟΕ ως Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που θα βοηθήσει το να πετύχουμε τα δύο τρίτα τη πλειοψηφία που χρειάζεται για να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. Πολλές σημαντικές χώρες ήδη έχουν πει δεν θα χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς τεχνολογικής υποστήριξης όπως η Κίνα παραδείγματος χάρη. Δεν θα χρειαστούν λοιπόν τεχνολογική τεχνική υποστήριξη για να εφαρμόσουν ε, τη συμφωνία και υπάρχουν και κάποιες διτάξει που είναι δεσμευτικέ, που αφορούν ε, τις οικονομικές ε, συναλλαγέ, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, εισαγωγέ εξαγωγέ, διακανονισμοί γύρω από αυτά τα θέματα που έχουν σκοπό τη μείωση ενό στόχου και στόχο αυτό είναι η μείωση τη διαφορά στο παγκόσμιο εμπόριο. Ε, ώστε να υπάρξει, μια, ε, μεγαλύτερη διαφάνεια στην παγκόσμια αγορά. Επίσης θα μειωθεί ο χρόνος ε, που χρειάζεται για τις συναλλαγές και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα, σύστημα παρακολούθησης των ροών. θα έχουμε διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για ένα πιστωρό ελεύθερο και πιο ασφαλές ε, διευθυντές σύστημα εμπορίου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να επικυρώσουμε ε, αυτή τη συμφωνία σε λογικό χρονικό διάστημα. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε μια έκθεση που θα είναι βασισμένη στη συνένεση και θα μπορέσουμε φυσικά να συνεισφέρουμε και με τη μορφή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία δυσκόλυνση εμπορίου είναι εξαιρετικά σημαντική σε επίπεδο παγκόσμιου εμπορίου, γιατί δεν έχουμε δει πολύ δραστηριότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει και μια έλλειψη συλλογική δράση και ω εκ τούτου αύξηση των διμερών ε, σχέσεων και επαφών. Είναι θετικό λοιπόν και το χαιρετίζουμε ως νέα εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντική και η δική μου κυβέρνηση επιθυμεί περισσότερα κονδύλια για την διεθνή ανάπτυξη και αυτό μαζί με την TFA είναι ένα άλλο μέσο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να ανοίξουμε το εμπόριο και να συνδράμουμε αυτές τις σχέσεις καθώς αναπτύσσονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Συγχαίρω και τον εισηγητή για τις συστάσεις του και ελπίζω η έγκριση να γίνει, η κύρωση μάλλον να γίνει με τα δύο τρίτα του ΠΟΕΠ το μέτρο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριο Μπούχνο. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο το οποίο μου άρεσε πολύ ομολογώ και αυτό που είναι σημαντικό για εμένα ότι ε, υπάρχει ένας ε, μοχλός για τη μείωση της δορδοκίας στους ε, τελωνικούς υπαλλήλους. Επίσης χαίρομαι που γίνεται λόγος για την ασφάλεια, για τα αναφορά στον Παλί και στην Ινδία. Θα ήθελα μια πιο σαφή διατύπωση και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο αυστηρή διατύπωση σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, I Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση που μας παρουσίασε. Δίνοντα έμφαση στο σύστημα παρακολούθησης και θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ ότι το, το γεγονό ότι θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική ώστε να υπάρχουν κοινέ λύσεις και προτάσεις για να βρούμε πολύπλευρους τρόπους οργάνωσης ε, του διεθνούς ε, εμπορίου παρά, παρά να επιμένουμε στις ε, διμερείς συμφωνίες. Και επίσης να τονίσω ότι είναι δύσκολο να πούμε όχι σε μια προσήγηση ήταν πάνω από 60% των χωρών, ειδικά οι χώρες από ε, τις ανεπτυγμένες χώρες έχουν συμφωνήσει ήδη. Φυσικά αυτό δείχνει ότι πρόκειται περί συμβασμού, αλλά παρόλα αυτά να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες που υπάρχουν από εμπειρογνώμενες και από τον ακαδημαϊκό χώρο και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. στο Μπαλί έγινε λόγος για τη συμπερίληψη του γύρου της Ντόχα και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην ε, προετοιμασία της νέας ε, υπουργικής ε, στο Ναϊρόμπι. Η πρώτη ανησυχία που θέλω να θίξω είναι ότι τα ωφέλη από τι ευκολύνσει ίσως υπερεκτιμώνται τόσο αναφορά στο έπος και στην απασχολησιμότητα. Οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν ζήτησαν να επενδυθούν εκατομμύριο με μορφή ε, κανονιστική και η δημιουργία υποδομών. Και αυτό με βάση την υπόσχεση ότι κάθε δολάριο που θα ε, επενδυθεί θα ε, αποδώσει 2 δολάρια και 87 σέντ σε ανάπτυξη αύξηση του ΑΕΠ. Μόλις μάθαμε ότι η Μεγάλη Βρετανία συμφώνησε και θέλει να επενδύσει περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. 400 εκατομμύρια έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης και άλλα πολλά εκατομμύρια από, από πολλά κράτη-μέλη του ΠΟΕΜ. Σε όλες τις εκθέσεις βλέπουμε ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα στην οικονομία. Άμα θυμάστε από την Αυτά και το, το Μεξικό, ε, κατάφερε να κερδίσει 7.000 επαγγέλματα στο μεταπητικό κλάδο, όμως έχασε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα. Οπότε υπήρξε μια αναδόμηση της εθνικής οικονομίας, που ε, είναι αποτέλεσμα αυτών των νέων συνεπειών αυτών των συμφωνιών. Υπήρξαν πολύ περίπλοκα θέματα με μπλοκή και τη μαφία των ναρκωτικών κτλ. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις εξελίξει και να μην ε, εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο στο εμπόριο. Δηλαδή το εντάξουμε το εμπόριο σε ένα πιο περίπλοκο ε, πλαίσιο. Να τονίσω επίσης ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την προσέγγιση μας με συνοδευτικά μέτρα που θα πρέπει να οδηγήσουν ε, να λάβουν υπόψη τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και τι αρνητικέ επιπτώσει που μπορεί να έχει αυτή η συμφωνία. Και τέλο, γίνονται βήματα για την αναδιοργάνωση τη οικονομία και υπάρχει μια, ένας προ ε, προς τις Κατά τη μεταβατική ε, περίοδο γίνονται, γίνονται και απόλυε στην αγορά εργασίας και υπάρχει ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα ε, προϊόντα, ειδικά στον τομέα της ε, γεωργία και στις αναπτυσσόμενες χώρε. Το Trade Facilitation Agreement του Μπαλί δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη όλο το σενάριο και έθιξε μονάχα κάποια παραδείγματα στην οικονομική αλυσίδα. Και έχουμε πάλι τα δικαίου εμπορίου προϊόντα τα οποία συνδέονται με μη δικές πρακτικές. Θα πρέπει να λάβουμε σε αυτά τα μικρά παραδείγματα. Θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα ε, στον εισηγητή και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία που θα αφήξει όλε αυτέ τι ανησυχίε ε, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ω Επιτροπή διεθνού Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σκαρατσότη, Επικεφαλή τη μονάδας τη Γενική Διεύθυνσης Εμπορίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη για τα καλά σα λόγια για αυτή τη συμφωνία. Ορισμένε παρατηρήσει αναφέρθηκαν από τα αξιότιμα μέλη σα. Πρώτον, για την ανάπτυξη θα παρασχεθούν κονδύλια, βεβαίω, Υπάρχουν και δέσμευση και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ πραγματικά απευθύνω έκκληση προς συντονισμό ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνδρομή ε, θα παρασχεθεί και επισήμω. Για τα ωφέλη. Υπάρχει νέα μελέτη του ΩΣΑ που μόλις ε, δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας Υπουργικής Συνόδου τον Ιούνιο για τα πιθανά ωφέλη και κόστη και προβλέπεται άνω του 15% για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι περισσότεροι τα έχουν συνδέσει όλα αυτά με το υπόλοιπο θεματολόγιο του ΠΟΕ. Βεβαίως είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως μια σημαντική πρόκληση σήμερα είναι ο ΠΟΕ να έχει αποτελέσματα στα κύρια στοιχεία και θέματα του θεματολογίου DDA ε, στο Ναϊρόμπι τον επόμενο Δεκέμβριο και αυτό είναι σημαντική πρόκληση και πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε του σύνεγγυς και με μεγάλη προσοχή όλες τις διαπραγματεύσεις και εξελίξεις μέχρι τα τέλη του χρόνου. Τώρα, για το τι ακριβώς είναι η συμφωνία ευκόλυνση του εμπορίου, τι έκανε και τι δεν έκανα. Δεν αφορά την περαιτέρω απελευθέρωση, αλλά το πώς θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε το επίπεδο απελευθέρωσης που έχει αποφασίσει ένα κράτος. Απελευθέρωση δηλαδή των δασμών και άλλων δομών που επιτρέπουν την απελευθέρωση. Το μέρος δηλαδή του ΠΟΕ παίρνει έτσι τα μέτρα που απαιτούνται για να συνδεθεί με τις παγκόσμιες ε, αλυσίδες αξιών. Δεν είναι μόνο για τις εισαγωγές, αφορά και τις εξαγωγές. Είναι κύριο στοιχείο για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξή σας. Παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε και για τις τρίτες χώρες για να στηρίξουν την πρωτοβουλία υπέρ της ε, έγκαιρη κύρωση τη συμφωνια έχουμε 66 μέλη του ΠΟΕ που ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης. Ε, όταν εμείς την κυρώσουμε θα μετρήσουμε ως 28 μέλη. Επομένω, ε, πλησιάζουμε το όριο των 108 χωρών για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η πρώτη συμφωνία του ΠΟΕ από το 1995 και μετά. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να μας οδηγήσει σε μια νέα επιτυχία το, στο Ναϊρόμπι του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής η συνάντηση στο Ναϊρόμπι. Πάμπλο. Ευχαριστώ. να τονίσω ακόμα μία φορά τη σημασία αυτής της συμφωνίας, τον πολυμερή του χαρακτήρα, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα θετικά και ευγενικά τους λόγια και να τονίσω τη σημασία να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν αυτό το δοσιέ, ούτω ώστε να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα στις υπόλοιπες χώρες και να πετύχουμε το όριο του των δύο τρίτων το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ για την ε, συνεργασία και συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ, Παύλο. Η καταληκτική ημερομηνία για την έκθεση αυτή θα είναι 23η Ιουνίου. Και τώρα. Περνάμε στο σημείο 6. Ο κύριος Μπορέλη δεν είναι Παρόλο ο ε, κύριο Μπικίν θα αναλάβει εκ μέρου του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματο του κυρίου Μπορέλη που δεν μπόρεσε να φύγει από την Ιταλία, θα ήθελα να σα καλώ να σκεφτούμε για την γνωμοδότηση αυτή. Να σα πω κάποιε ιδέε. Καταρχά, πριν πω στο περιεχόμενο, θα ήθελα να σταθώ μια στιγμή στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Η γνωμοδότηση που συζητάμε και που αύριο θα ψηφιστεί είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας ε, και χάρη στην προσπάθεια πολλών συναδέλφων της Επιτροπής. Οι διάφορες ιδέες ε, ήταν, μας εξυπηρέτησαν και αποτέλεσαν βάση αυτού του κειμένου που βλέπετε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λάγκε Μπούχνερ, Λάγκε Μάρτιν, Πατριτσέλο Ρούας και Σάκε για τις ιδέες τους. Αυτές οι ιδέες μου επιτρέπουν τώρα να, μετά από αυτά θα ήθελα να περάσω στα πολιτικά θέματα, που είναι πολύ σημαντικά για την έκθεση αυτή. Οι συνάδελφοι έδωσαν σημασία, και αυτό φάνηκε και από τις τροπολογίες, ε, στο θέμα της ε, επικουρικότητας που ξεπερνάει πολύ το πεδίο εφαρμογή αυτής της νομολογίας. Ο πρόεδρος Γιούνκερ πρόσφατα ε, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα με μία σειρά από πρωτοβουλίε. Ε, πιο γνωστή είναι το Better Regulation, ούτω ώστε να έχουμε μια καλύτερη ε, εφαρμογή της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών. Έχουμε λοιπόν το θέμα της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις που θα εξυπηρετούν και θα είναι πιο κοντά στους πολίτες μας. Μία γενική έτσι, και υπερτροφική Ευρώπη απομακρύνει τους πολίτες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό ελπίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή θα βοηθήσει στη συζήτηση που είναι εξελίξη για το better regulation. Όπως ξέρετε, το θέμα της επικουρικότητας δεν ε, εξαρτλείται στο πού θα παρέμβουμε, δηλαδή στο εθνικό ή στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, για τις ευρωπαϊκές ας πούμε, συνθήκες όπως το TTIP. Είναι ε, αφορά το άρθρο 1, αυτό που μιλάει για τις μεικτές συμφωνίες ή για περιπτώσεις όπου και τα εθνικά κράτη εκφράζονται. Δείτε μια σημαντική έμφαση στο θέμα της διαφάνειας και της λογοδοσία στι διαπραγματεύσει. Εδώ πολλέ πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Συχνά θέτουν το ερώτημα, αλλά δεν το ακούνε πολύ, ε, ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες για τι διαπραγματεύσεις πάνω στο TTIP, Φερρυπίν. Ε, θέλουμε ε, διαφάνεια ε, και το θέμα αυτό είναι οριζόντιο. Αφορά τους, όλους τους επιτρόπους και όλα τα χαρτοφυλακιά τους. Το δεύτερο και τρίτο σημείο αφορούν την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική και το θέμα του SDS, του ISDS, την επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτών. Ε, αυτό αφορά και τις αρμοδιότητες της Ένωσης και τις εθνικές αρμοδιότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια για τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ή ε, τον κίνδυνο που έχει το ISDS για τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Η, πολιτική, η οικονομική πολιτική εσφαλμένα θεωρείται ότι αφορά μόνο την επικουρικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το τέταρτο σημείο είναι το θέμα της μακροοικονομικής βοήθειας και αναφέρεται σε μεγαλύτερους ελέγχου ε, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Δεν θέλουμε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί ε, μόνο επικουρικά, χωρίς όρια. Ε, με χαρά είδα ότι υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ των πολιτικών ομάδων που θέλουν μεγαλύτερο έλεγχο για να αντιμετωπίσουμε απάτες και διαφθορά, καθώς και μεγαλύτερο συντονισμό με άλλα εργαλεία της ε, εξωτερικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, γίνεται ε, αναφορά στις ε, μελέτες αντικτύπου που συχνά χρησιμοποιείται λάθος. Ε, θα θέλαμε πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει να γίνονται αυτέ οι μελέτε αντικτύπου και όχι αφού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Ε, για να μην γίνονται μόνο εκ των υστέρων αξιολο... ε, αντικτύπου που θα είναι επισφαλής. Το σημείο 6 αφορά την εμπλοκή των πολιτών ε, στη λειτουργία των ε, επιχειρήσεων, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη λήψη των αποφάσεων στα θέματα εμπορικής πολιτικής. Ε, ο διάλογος και η δημοκρατική εμπλοκή είναι πολύ σημαντικά θέματα και να περιοριστούμε και δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στα τυπικά θέματα. Πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο κατόφλι ε, για τη συμμετοχή των πολιτών, τόσο ώστε να αξιολογούμε εάν η δημόσια διαβούλευση ήταν αποτελεσματική ή όχι. Θα κλείσω ε, τονίζοντα την πολιτική σημασία του περιεχομένου αυτή τη έκθεση και τη μεθόδου που ακολουθήσαμε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τον David Μπορέλη και του συναδέλφου που συνεισέφεραν στην, ε, στο κείμενο αυτό. Ε, δεν μιλάμε μόνο για αφηρημένε έννοιε, αλλά μιλάμε για πολύ λεπτά θέματα που στο μέλλον θα επηρεάσουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάτε ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, αλληλεπιδρούν με τους πολίτες τους. Ελπίζω να υπάρχει μεγάλη και ευρεία και πλατιά συνένεση για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν σχόλια, επιθυμία να πάρουν το λόγο σκιώδες ηγετές. Να σχολιάσουν και τις τροπολογίες. Παρακαλώ. κάποιες παρατηρήσεις την κυρία Καρίν, η οποία δεν είναι εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το άρθρο του. Οκ, okay, έχει να κάνει με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Να το ευχαριστήσω για, το, για την έκθεση, αλλά και που έλαβε υπόψη κάποιε τι ανησυχίε των μελών. Υπάρχει μεγάλη στενή που φαίνεται από, ε, από του συμβασμού. Και οι δύο αυτέ οι έννοιε θα είναι πολύ σημαντικέ στην νομοθετική διαδικασία. Υπάρχουν δύο βασικά σημεία που είναι σημαντικά για την δικιά μου ομάδα. Αφορά το ένα τη μελέτη αντικτύπου και ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκή Ένωση Όσον αφορά τις ε, μελέτες αντικτύπου, είναι πολύ σημαντικές γιατί έχουν αναφορές σε δεδομένα και αντικατοπτρίζουν ε, αποφάσεις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί. Και ήταν πάντα πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες ε, για την εφαρμογή της πολιτικής και έχουν εδώ δείξει πολλές ε, ωφελήσει την αύξηση των ε, κερδών από το εμπόριο, όπως παραδείγματο χάρη η συμφωνία με την Κορέα μας έχει δείξει ότι, ότι αυτά που εκτιμήθηκαν και αντίθετα με κάποιες ανησυχητικέ ε, προειδοποιήσει ότι ήταν καλή συμφωνία για την οικονομία και όσον αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλιο ε, η Κομισιόν θέλει να παραπέμψει στο ECA Τώρα που με μελετάμε λεπτομερώ πώ θα αυξήσουμε ε, την, το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και της, ε, του Πρόεδρου τη Επιτροπής. Ευχαριστώ. Um Αυτή είναι μια έκθεση που συζητήθηκε στην Επιτροπή επί Δικαιοσύνης και πέρα από το θέμα της επικουρικότητας και την κοινή πολιτική ότι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία υπάρχουν συγκεκριμένες ε, εξαιρέσεις που αφορά τη μακροοικονομική υποστήριξη τρίτων χωρών αυτό αναφέρεται στο άρθρο 112 και να ευχηθούμε ότι ε, η έκθεση του κ. Μπορέλη θα λάβει απόψε αυτές τις δύο πτυχές και είναι γεγονό ότι η πλειοψηφία ε, θα δεχτεί τις τροπολογίες που έχει προτείνει ο κ. Μπορέλη. Υπάρχουν έξι συμβαστικές προτάσεις, αλλά η τροπολογία 22 για το εδάφιο 5 δεν λήφθηκε υπόψη επιπαρκώ στην συμβαστική λύση 5 και γι' αυτό υπάρχει, μια ε, εναλλακτική πρόταση η οποία αντιμετωπίζει πιο λογικά αυτό το θέμα για την εκ των ε, εκτίμηση, εκ των προτέρων εκτίμηση. και που θα είναι πολύ επαφέλε τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη συμβαστική πρόταση 6, υπάρχουν επιφυλάξεις σε αυτή την πρόταση. Ε, να υπάρξουν κάποια ελάχιστα κριτήρια, δηλαδή κριτήρια ε, πρόσβασης όταν θα αφορά συγκεκριμένες ομάδες πολιτών ή κρατών, αλλά κατά τα άλλα υποστηρίζουμε πολύ το πολύ καλό έργο και αυτό που είναι σημαντικό να υπάρξει, είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους, ε, στα θεσμικά όργανα και να προσπαθήσουμε επίση να υπερβούμε ε, τα ελληνικά εμπόδια, να έχουμε μια πιο δίκαιο, ένα πιο δίκαιο και πιο ισορροπημένο εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot. Herr Κύριε Σούστα, ο Λάιχτ Φρίντ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και γι' αυτό με παρακάλεσε να θίξω κάποια σημεία για την έκθεση για την αναλογικότητα και την επικουρικότητα του 2013. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, την καλή συνεργασία καταφέραμε να καταλήξουμε σε έξι συμβαστικέ λύσει. Είναι αναγκαίο από ό,τι φαίνεται να διαχωρίσουμε ε, τις αρμοδιότητες μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτέ τι συμφωνίε και να σεβαστούμε και τι δύο αυτέ ε, αρχέ. Στι διεθνεί διαπραγματεύσει. σε μόνο θετικά ε, αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε όταν σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες δεν ενεργεί μονομερός κάθε κράτος μέλος ε, και όλα αυτά φυσικά συμπεριλαμβάνονται και στην συνθήκη της Λισαβόνας. Βασικό αίτημα είναι κάποια μέλη να ε, αφήσουν την ε, θέση μπλόκου που κατέχουν Όλα τα κράτη-μέλη ε, είναι συμβαλόμενα μέρη σε αυτή τη συμφωνία. Και αυτό για να αποφύγουμε την, ε, τις στρεβλώσεις στην αγορά. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερος διάλογος και εμπλοκή της κοινωνία των πολιτών στην διαδικασία ε, αποφάσεων, λήψη αποφάσεων. Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι που θα ήθελα να πάρουν το λόγο και γι' αυτό το λόγο ολοκληρώνουμε τη συζήτηση ε, για την ε, έκθεση και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο της μερικής διάταξης 10. Πρωτού μπούμε στο σημείο 1. Θα ήθελα να σας πω ότι οι συντονιστές χθες αποφάσισαν να έχουμε μια νέα συνεδρία στις 29 Ιουνίου από τις 3 μέχρι τις 4.30 θα γίνει η συνεδρίαση συντονιστών την 29 Ιουνίου και μετά θα ακολουθήσει ε, συζήτηση για τις 116 προτάσεις τροπολογίας για το τίτλο από την Ολομέλεια και μετά θα γίνει ψηφοφορία εκτός μικροφώνου. Επαναλαμβάνω, 29 Ιουνίου. Νέα συνεδρίαση στις 3 ώρα το απόγευμα με τους συντονιστές μέχρι τις 4.30. Στις 4.30 θα ακολουθήσει συζήτηση για τις 116 ε, προτάσεις τροπολογίας από την Ολομέλεια και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε αν θα εγκριθούν αυτές τις τροπολογίες Όταν ε, πέντε μέλη της Επιτροπής είναι υπέρ, τότε παραμένουν τροπολογίες. Όμως σίγουρα θα συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το θέμα. 29 Ιουνίου λοιπόν. Συνεδρία συντονιστών μέχρι τις 4.30 και στη συνέχεια συζήτηση επί του και ψηφοφορία. Κατά δεύτερον. Και πάλι εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Σας παρα... παρακαλέσω ε, στην ψηφοφορία να μην ε, ε λάβουν η βοηθή να δούμε πραγματικά ποιος από τα μέλη είναι όντως παρόν. Να ξεκινήσουμε με τις κάρτες για να δούμε πόσοι είστε παρόντες. Άρχεται η ψηφοφορία.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 θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. πρώτα για το θέμα τη ψηφοφορία, συγγνώμη. Πριν δούμε τα πρακτικά, μπορούμε να δούμε τι ψηφίζουμε. Δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζουμε. Uh, Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα, παρακαλώ. Πριν κάνουμε τη δοκιμή της ψηφοφορίας, μπορούμε να μάθουμε τι θα ψηφίσουμε, να συζητήσουμε και τι θα ψηφίσουμε. Ich bin ein bisschen Έχω μείνει έκπληκτος, ομολογώ. Έχουμε τη σειρά της οφορίας, έχουμε το σημείο 10. Μίλησαμε ήδη για την έκθεση για την επικουρικότητα και μετά ξεκινάμε με τα επόμενα σημεία. Αυτή είναι η σειρά της ψηφοφορία όπως την έχετε στην ημερήσια διάταξη, κυρία Ρένα. Για το δεύτερο σημείο της ψηφοφορία, τον τρίλογο δηλαδή, για τα μεταλλεύματα από περιοχές σύγκρουση. Εκπλήσωμε που βλέπω ότι ψηφίζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ψηφίζουμε το να ξεκινήσει ο τριμερή διάλογο και δεύτερον ψηφίζουμε τη σύνθεση τη ομάδα που θα πάει στον τριμερή διάλογο. Δεν αμφισβητώ το να ψηφίσουμε τη σύνθεση της ομάδας που θα πάει στον τριμερή διάλογο, γιατί αυτό ήθελε και η Ολομέλεια, αλλά όμω βρίσκω ότι είναι ιδιάζον που θα πρέπει να ψηφίσουμε στην ίντα αυτό που ψηφίστηκε ήδη στην Ολομέλεια. Δηλαδή ότι μπαίνουμε δηλαδή σε τριμερή διάλογο, ξεκινάει ο τριμερής διάλογο. Εσεί, πρόεδρος, πρόεδρε που ζητήσατε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, το να ξεκινήσει ο τριμερή διάλογο. Είναι φυσιολογικό δηλαδή να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε δύο φορές, μία φορά στην Ολομέλεια και μία φορά στην Επιτροπή. Το να ξεκινήσει ο τριμμένος διάλογος. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω. Γιατί εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τη διαδικασία. Και μάλιστα αμφισβητώ το να ψηφίσουμε δεύτερη φορά εδώ στην Επιτροπή ΙΝΤΑ το, το θέμα της εκκίνησης του τριμμένου διαλόγου. Κυρία Ρένα, για να είμαι ξεκάθαρο, στην Ολομέλεια αποφασίσαμε την παραπομπή και πάλι στην Επιτροπή για το θέμα του ε, τριμερούς διαλόγου και μετά ε, κάναμε μια στα άρθρα 72-2 και 72.3 του αστικού κανονισμού που κάνει λόγο για την ε, ε, απόφαση με πλειοψηφία στην Επιτροπή για την έναρξη του διμερούς διαλόγου και ενεργώ φυσικά σύμφωνα με τον ε, εσωτερικό κανονισμό Ρώτησαμε και την νομική υπηρεσία. Είναι εδώ η νομική υπηρεσία μάλλον για να μας το παρουσιάσει λίγο πιο μέρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Θα ήθελα να απαντήσω στην παρέμβαση της κυρίας Αρένα. Πράγματι θεωρώ ότι η Ολομέλεια ξαναέστειλε το θέμα στην Επιτροπή, όμως δεν μπορεί η Ολομέλεια βάσει του 73 παράγραφος 2 του Οστρικού Κανονισμού να αποφασίσει. Δηλαδή, κατά πόσο η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα έπρεπε να ξεκινήσει τριμερή διάλογο. Αυτή η απόφαση εναπόκειται στην Επιτροπή σα και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κανόνα ψηφοφορία, δηλαδή απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να αποφασίσετε εάν θέλετε ε, να εισέλθετε σε διαπραγματεύσει ή όχι. Δεν είναι δηλαδή απόφαση της Ολομέλειας, είναι απόφαση της Επιτροπής, γιατί παρέπεμψε η οχι δεν ειναι δηλαδη αποφαση της ολομέλεια, ειναι αποφαση της επιτροπης γιατι παρεπεμψε η ολομελεια στην Επιτροπή ε, την απόφαση αυτή. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα προτείνατε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαντό θέλει να πάρει το λόγο και δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε με διάλογο επί του θέματος αυτού. Κι όμως είναι ιδιαίτερη αυτή η ερμηνεία των όσων συνέβησαν στην Ολομέλεια. Όλοι ήμασταν εκεί. Πράγματι τα όσα ψηφίστηκαν, τι ήταν δηλαδή, τι ψηφίστηκε η έναρξη των διαπραγματεύσεων και επί της ουσίας μας λένε ότι η Ολομέλεια δεν ε, υπερισχύει, δεν έχει την κυρίαρχη θέση. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Όταν αποφασίζει η Ολομέλεια, αποφασίζει ότι μετά εντάξει το να ψηφίσουμε τη σύνθεση και το καθεξής αυτό είναι απολύτως λογικό. Όμως η Ολομέλεια αποφάσισε να εισέλθουμε σε διαπραγματεύσεις και μετά υπάρχει μια ασαφής ερμηνεία ε, της ε, κυρίαρχης αυτής ε, ψήφου τη Ολομέλειας. Κύριος Κάσπαρ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω για δύο θέματα. Το ένα που ανέφερα και χθε στη συνεδρίαση των συντονιστών, θα το πω και ανοιχτά, έχει να κάνει με τον τρόπο και τη μορφή τη συνεργασία. Στην τελευταία περίοδο είχαμε πάντα τη συμφωνία για το αν θα παραπέμπονται εκ νέου κφάκελοι από την Ολομέλεια στην Επιτροπή. Αυτό που έγινε στην Ολομέλεια ήταν κάτι που έγινε πρώτη φορά. Η δικιά μου ομάδα ενημερώθηκε, κάποιοι άλλοι ομάδες δεν ενημερώθηκαν και δεν είχαν σχετικά σχέδια και φυσικά σύμφωνα με τον ε, ιστορικό κανονισμό ε, και πάλι ε, στην Επιτροπή το θέμα. Και τώρα, επιπλέον, σαν να μην έφτανε αυτό, θέλουν οι συνάδελφοι να συζητήσουν ε, για ε, τον εσωτερικό κανονισμό, κάτι που είναι όμω πολύ σαφές. Και παρακαλώ να ψηφίσουμε εδώ, σύμφωνα με τον κανονισμό, για να μην ξεκινήσουμε διαλόγους. Φυσικά υπήρξε που δεν ήταν και τόσο σαφέ στην Ολομέλεια. Τώρα όμω είναι πιο, ε, μπορούν να καταστούν πιο σαφή αυτά με βάση τα άθρα του εσωτερικού κανονισμού. Α ακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδικασία για να μην καθυστερήσουμε άλλο με συζήτηση επί του θέματο. Ε, λοιπόν, για να είμαστε σαφεί, λέει ο Πρόεδρο, η συζήτηση στην ε, Ολομέλεια αφορούσε το άρθρο 62.1 του ιστορικού κανονισμού και φυσικά δεν ε, έγινε κάτι, ε, δεν έγινε κάποιο κόλπο εκεί. Κάναμε ένα διάλειμμα και συνέχεια η Ολομέλη αποφάσισε να παραπευθεί το θέμα στην Επιτροπή το θέμα της συμμετοχής στον τριμερή ε, διάλογο και έτσι λοιπόν σύμφωνα με τη δικασία θα πρέπει να αποφασίσουμε για αυτό το θέμα εδώ. Είναι πάρα πολύ σαφές, είναι πολύ σαφής ο εσωτερικός κανονισμός και θα τον τηρήσω. Είναι κάτι που πρέπει να το αναμένετε από εμένα και είναι και κάτι που θα ήθελα και να το εγγυηθώ. Αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν. Λοιπόν, προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για την ε, έκθεση για την επικουρικότητα του κυρίου Μπορέλη. Και περνάμε στην ψηφοφορία για την ε, ε, πρώτη τη ευρωβουλευτική. Ένα. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχέ. Και αυτή εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογία 6. υπέρ και κατά. Πιστεύω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Excuse me. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Η ερμηνεία λέει συμβιβασμό 6. Εννοούσατε τροπολογία 6. Τροπολογία 6 ή συμβιβασμό 6. Είναι καλή, σωστή αυτή η διευκρίνηση. Είναι η τροπολογία 6 του κυρίου Λάιχφριτς. Abstimmung ist eröffnet. Άρχεται η ψηφοφορία και κλείνει και εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογίες 7. Ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κακά, κατά, αποχές και αυτή εγκρίνεται. Πρώτες τροπολογίες 9. Και αυτή εγκρίνεται. Πρόταση συμβιβασμού 3. Ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά. Αποχές και αυτή εγκρίνεται. Πρόταση τροπολογίας 10. Καταπίπτει. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές και αυτή δεν εγκρίνεται. Πρώτα συμβασμού 4 υπέρ κατά και αποχές και αυτή εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογίας 16. Καταπίπτει. Πρώτα συμβασμού 5 υπέρ κατά και αποχές. Ας το ελέγξουμε λίγο καλύτερα. Πρώτα συμβασμού 5 άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Δεν εγκρίνεται. Πρόταση συμβασμού 5α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρόταση τροπολογίας 23. Δεν εγκρίνεται Πρώτα συμβασμού 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Και αυτή δεν εγκρίνεται. Πρόταση τροπολογίας 26. Εγκρίνεται. Πρόταση τροπολογίας 28. Ε, ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την πρόταση τροπολογία 28. Έχει κλείσει η ψηφοφορία και δεν εγκρίνεται και περνάμε στην ε, ψηφοφορία επί του συνόλου των τροπολογιών ε, το του σχεδίου έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχει κλείσει η ψηφοφορία. Με 30 ψήφους εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπορέλη. Jetzt kommen wir Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τη γεωγραφική ένδειξη σε μη προϊόντα. Πρόταση συμβιβασμού 4. Ξεκινάμε με αυτή την πρόταση. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτα συμβασμού 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην πρόταση τροπολογίας 10. Δεν εγκρίνεται. Πρόταση τροπολογίας 11. Υπέρ κατά και αποχές εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογία 12. Εγκρίνεται. Πρώτα συμβασμού 2. Υπέρ. Κατά. Και αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογία 19. Εγκρίνεται. Πρώτο συμβασμού 3. Εγκρίνεται. Πρώτο συμβασμού 6. υπέρκατα και εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. υπέρκατα και αποχέ δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογία 34. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Και αυτή δεν εγκρίνεται. Πρώτος τροπολογίας 36, υπέρ, κατά και αποχές. Δεν εγκρίνεται. Πρώτες συμβασμού 5, μια παρατήρηση. Πήξε το ζήτημα αν, κατα... αν καταπίπτει μαζί με αυτήν και η πρόταση τροπολογίας 39 η οποία τελικά ε, καταπίπτει αν εγκριθεί η πρώτα συμβασμού 5. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτα συμβασμού 7. Υπέρ κατά. Και αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά δεν εγκρίνεται. Πρώτα τροπολογία 44. Δεν εγκρίνεται. 45. Υπέρ, κατά και αποχές. Δεν εγκρίνεται. Πρώτες τροπολογία 46. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Επίσης δεν εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την ε, αλλαγή της ε, ε, επί του συνόλου της έκθεσης έχει κλείσει ψηφοφορία και πάλι με 30 ψήφους εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Μόσκα που σήμερα δεν παραβρίσκεται σημείο 13 ψηφορία για την έναρξη του τριμερούς διαλόγου και τη σύνθεση της αντιπροσωπείας. Θα ήθελα μια μικρή διευκρίνηση. Υπενθυμίζω ότι η Ολομέλεια ψήφισε να πάμε σε τριμερή διάλογο. Εάν μετά τη σημερινή ψηφοφορία εδώ στην ε, Επιτροπή ψηφίσουμε διαφορετικά από ότι η Ολομέλεια. Θα ήθελα μια νομική γνώμη για τη θέση που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή έχουμε 751 βουλευτές που ψήφισαν στην Ολομέλεια που είπαν να πάμε στον τριμερή διάλογο. Τώρα δηλαδή οι 40 βουλευτές ε, της ΙΝΤΑ έχουν περισσότερη ισχύ από τους 751 της Ολομέλειας. Τι θα γίνει τελικά, θα ήθελα επίσημη θέση της ε, νομικής υπηρεσίας για αυτό το ζήτημα. Wir sind in der Στον ιστορικό κανονισμό δεν δεσμευόμαστε για εναλλακτικέ λύσει. Θα ρωτήσουμε του συντονιστέ για το πώ θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ, αλλά αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ε, τη ε, απόφαση τη ομάδα συντονιστών. Λοιπόν, Περνάμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια δημοκρατική, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Ότι θεωρώ ότι η παρατήρησή σας ότι αυτό είναι θέμα ε, των συντονιστών, αυτό με ξενίζει πρέπει να πω. Στην αρχή της θητείας λάβαμε κάποιες διαδικαστικές αποφάσεις ε, με τους ε, συντονιστές και να αποφασίσουμε και το πώς θα προχωρήσουμε. Και στον ιστορικό κανονισμό δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ε, ρυθμίσεις. Ναι, υπάρχει δημοκρατική βάση και υπάρχει και συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει σύμφωνα με τον στήριο κανονισμό να αποφασίσουμε σήμερα αν θα προχωρήσουμε στον τιμερή διάλογο και ποιο θα ηγηθεί τη ε, ομάδα των αντιπραγματεύσεων. Κύριε Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όμω. Εντάξει, εγώ δεν ε, είμαι θαμώνα εδώ τη Επιτροπή, όμω είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα γιατί η ψηφοφορία στην ομέλεια ήταν σαφής Θυμάστε εσείς, δηλαδή ψηφίσαμε να περάσουμε στον μερή διάλογο. Τώρα αμφισβητούμε ουσιαστικά μία ε, απόφαση της ε, Ολομέλειας, όχι μόνο εδώ ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά θα μπορούσε αυτό το θέμα να τεθεί ε, σε συμφορία στους συντονιστές, ενώ ένας μόνο νομικός μας πήρε μία θέση. Γιατί αν ε, ρωτήσουμε δύο νομικούς, θα έχουμε τρεις γνώμες. Εδώ εμπιστευόμαστε μόνο έναν νομικό για να αντιστρέψουμε ενδεχομένω ε, την ε, απόφαση Ολομέλεια. Κύριε Γιασπάρη, είναι απαράδεκτο εσεί να ερμηνεύετε τα όσα συμβαίνουν στην Ολομέλεια επειδή δεν σα άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σαφέ. Και είναι πολύ σοβαρό. Για πρώτη φορά, εγώ δεν έχω προηγούμενο στην ιστορία του Κοινοβουλίου να αμφισβητούμε την ψηφοφορία, το τελικό αποτέλεσμα στην Ολομέλεια, γιατί δεν συμφωνούμε με το αποτέλεσμα. Ich glaube, es hilft wirklich. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει να διαβάσουμε λίγο τον ιστορικό κανονισμό. Συμπτωματικά τον έχω μαζί μου. Das heißt 3. Άρθρο 73.3 και λέει και 73.2 του ιστορικού κανονισμού. κάνει λόγο για ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Γίνονται αποδεκτές οι διαπραγματεύσεις μόνο όταν η αρμόδια επιτροπή με πλειοψηφία των μελών εγκρίνει την ε, έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων. Όταν εγκρίνει δηλαδή η αρμόδια επιτροπή διαβάζουμε τον κανονισμό που λέει ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ δεν μπορεί να ε, πάει στον τριμερή διάλογο εάν δεν έχει την ε, σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών. Αυτό είναι σωστό. Όμως τι συμβαίνει όταν η Ολομέλεια έχει ψηφίσει και αποφασίσει πριν από την Επιτροπή. Αυτό συνέβη. Πριν από την Επιτροπή Ίντα αποφασίσαμε ήδη να πάμε στην μέρη διάλογο. Εσεί διαβάζετε το άρθρο του ιστορικού κανονισμού που λέει τι πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο τη Επιτροπή. Όταν δεν υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου. Όμω σήμερα υπάρχει θέση 751 βουλευτών και εσεί μου διαβάζετε ένα άρθρο του εθνικού κανονισμού που λέει τι κάνουμε όταν δεν έχουμε πάει στην Ολομέλεια. Όμω εμεί πήγαμε στην Ολομέλεια. Και τι είπε η Ολομέλεια. Έχουμε ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο. Επομένω η Επιτροπή μα δεν λαμβάνει πλέον θέση επί του ζητήματο. Απλώ αποφασίζει την τελική σύνθεση τη ομάδα, οργανώνουμε ε, τον τριμερή διάλογο και το καθεξή. Όμω είπατε και εσεί ότι δεν προβλέπει το ο ιστορικό κανονισμό να έχουν αποφασίσει κάτι στην Ολομέλεια που θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από την Επιτροπή. Και εσεί λέτε ότι οι συντονιστέ μάλιστα θα το αποφασίσουν. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Υπήρξε δημοκρατική απόφαση στο Κοινοβούλιο και εσείς θα περιορίσετε ε, την απόφαση αυτή σε επίπεδο συντονιστών. Είναι απαράδεκτο. Ζητώ να πάει στη διάσκεψη των Προέδρων το ζήτημα και να αποφασιστεί εκεί. Λοιπόν, κυρία Αρένα, δεν είπα ότι... Ε, είπα ότι θα αποφασίσει η Επιτροπή και θα πρέπει να το τηρήσουμε αυτό. Μόνο ότι υπάρχει αρνητική ψήφος τότε Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό κύριε Κασπάρη. Λοιπόν, δέχτηκα προσωπική επίθεση, δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν και θέλω να σας θυμίσω ότι στην Ολομέλεια αναφέρθηκε ο πρόεδρο σε ένα άρθρο του ιστορικού μα κανονισμού και σύμφωνα με αυτό το άρθρο ζήτησε να γίνει παραπομπή και πάλι στην Επιτροπή. Αυτό ήταν το αίτημα και αν κατάλαβα καλά δήλωσε την πρόθεση ότι θα πρέπει ως Επιτροπή να ξεκινήσουμε το θέμα σε συντριμερή διάλογο. Όμως η δημοκρατία δεν αφορά την δύναμη του ισχυρού, αλλά τη δύναμη του δικαίου, τη ισχύ του δικαίου. Και γι' αυτό το λόγο παραπέμφθηκε το θέμα στην Επιτροπή. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το αίτημα. Έχω τα πρακτικά τη ε, ολομέλεια. Σύμφωνα με το 61 παράγραφος 2 Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια και στη συνέχεια λήφθηκε υπόψη και ο εσωτερικό κανονισμό και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρήσουμε κι εμείς ε, τη διδάξη του εσωτερικού κανονισμού. Ο εσωτερικό κανονισμό που διαβάζεται υφίσταται αδιαμφισβήτητα. Όμω, θα ήθελα να πείτε στην προσοχή των συναδέλφων στο γεγονό ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντο όλες οι δεσμεύσει και αποφάσει για την έναρξη τριμερών διαλόγων γίνονται στην Ολομέλεια, όχι στην Επιτροπή. Είναι θέμα ουσία ο τρόπος δηλαδή η μέθοδος λειτουργίας που ακολουθούν οι επιμέρους επιτροπές. Άκουσα τα όσα είπε ο κ. Κασπάρη για μια ερμηνεία των όσων έχουν συμβεί, όμως εάν ο κ. Κασπάρη ψήφισε για να δούμε εάν θα ε, ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει ή όχι, σίγουρα οι υπόλοιποι 751 ε, ψήφισαν ξεκάθαρα. Όχι δηλαδή για να στείλουν το ζήτημα στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα εδώ. Ich lasse jetzt noch... Λοιπόν, ας περάσουν ε, και τα μέλη της άλλες πολιτικές ομάδες, κύριε Σούλτ. διάβασε ο κ. Κασπάρη τα πρακτικά και ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο. Το ψήφισε η Ολομέλεια και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά της ε, Ολομέλειας για έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συζητήσαμε τη περαιτέρω συνεργασία ε, για το θέμα αυτό χθε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Κύριε Μπεγκίν. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία Αρένα, τον κύριο Σόλτ, με τον κύριο Ζαντό. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι στην Ολομέλεια ψηφίσαμε για να παραπεμφθεί το θέμα, η συζήτηση δηλαδή, στον τριμερή διάλογο, κατευθείαν. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Τώρα θέλουμε να ξαναερμηνεύσουμε τους κανόνες, μόνο για να ευχαριστήσουμε κάποιους πολιτικούς οι οποίοι είναι πολιτικοί πολιτικάντιδες, με πι μικρό, όχι με πι κεφαλαίο. Αγαπητέ συνάδελφοι, δεν πρέπει να βιαστούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχουμε πιέσει και το Συμβουλίο είναι σε μια φάση ε, συμφώνιων και επειδή έχουμε στι 29 μια νέα συνεδρίαση θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ψηφοφορία στις 29 του μήνα ώστε να υπάρξει νομική σαφήνεια να είμαστε σίγουροι δηλαδή για την νομική ισχύ για το αν πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο αυτό στην Επιτροπή Κυρία Σάρκε. Σάκε. Κύριε Πρόεδρε. Απέχουμε πολύ από το να ψηφίσουμε μία έκθεση ή να μπούμε σε ένα τεμερη διάλογο για μια έκθεση που έχει ως στόχο την εξέβρεση λύσεων για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τώρα βλέπουμε ότι Περνάμε σε μικροπολιτικές προσεγγίσεις, ακολουθεί ο καθένας ε, περίεργες ε, τακτικές ε, για να περάσει το δικό του και καλώ του συναδέλφου που δεν έχουν πάει σε τριμερεί διαλόγου στο παρελθόν να δουν πώ ακριβώ αυτή του συστάση αποδυναμώνει τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Τώρα το αφήνω στη δική σα διακριτική ευχαίρεια για το πώ θεωρείτε εσεί ότι πρέπει να εφαρμόσουμε του κανόνε, ούτω ώστε να είναι ε, δίκαιοι οι κανόνε του παιχνιδιού για όλου. Αν εσεί θεωρείτε ότι πρέπει να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία, δική σα είναι η απόφαση, όμω δεν ξέρω τι ακριβώ περαιτέρω σαφήνεια χρειαζόμαστε. Και ελπίζω αυτά και είμαι σίγουρη μάλλον ότι τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα θα μας ε, απομακρύνουν ακόμα περισσότερο από τον τελικό στόχο που είναι να ρυθμίσουμε ακριβώ το ζήτημα της, ε, των μεταλλευμάτων από ε, Έμα. Έχουμε την μερική διάταξη, το συζήτησαμε χθε το θέμα. Εγώ δεν έχω λόγο να αναβάλω αυτή την ε, τροπολογία και να αμφισβητήσω το λόγο για τον οποίο συμπεριλήφθη στην μερισία διάταξη. Θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Πρόεδρε, έτσι που όπως εξελίσσεται η συζήτηση, άκου άκουσα την κυρία Σάκη να μας λέει αντίδες, ενώ το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ε, πήρε απόφαση. Πού είναι η μικροπολιτική όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση της, ε, στην Ολομέλεια κυκλοφόρησε μια νομική, ένα νομικό σημείωμα άτυπο. Ίσως η έκθεση της 29ης Ιουνίου να μας επιτρέψει να έχουμε και μια νομική γνωμοδότηση ε, πιο σοβαρή και ένα επίσημο, μια επίσημη νομική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό της ψηφοφορίας. Πρόεδρε, δεν θέλω να χρονοτριβήσουμε, αλλά είμαι εισηγητής παρόλα αυτά. Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Είχαμε σαφή ψηφοφορία στην Ολομέλεια και έχουμε και τον εσωτερικό κανονισμό. Κανένα από του αξιότιμους συναδέλφου, δεν θα πρότεινε να ψηφίσουμε και για τον εσωτερικό κανονισμό, φαντάζομαι. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνάδελφο, το πρόβλημα που έχω είναι αυτό που είπε η Μαρίτη Σάκε αν θέλουμε να δούμε με σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα, τότε δεν έχει πραγματικά νόημα να μπούμε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις και ε, να ξεφύγουμε ουσιαστικά από την ουσία του πράγματος και να συζητήσουμε αυτές τις πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, έχουμε τη συνεδρία στις 29 Ιουνίου. αναβάλουμε για τότε την ψηφοφορία ώστε να είμαστε ξεκάθαροι. Χθε στη συνεδρία στο Συντονιστό, το συζητήσαμε αυτό το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχουμε μόνο μία ευκαιρία να λάβουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ως κοινοβούλιο όταν αν θέλουμε να εργαστούμε αν θελουμε να εργαστουμε επικοδομητικά με τους άλλους. Επιπλέον, αν δεν ε, Λειτουργήσουμε ως εξής θα μπορούσαμε να έχουμε μια ε, λογική τοποθέτηση και έναντι των υπόλοιπων ε, θεσμικών οργάνων. 29 Ιουνίου λοιπόν αναβάλλεται για τότε ψηφοφορία.